πολιτική της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης ώστε να λήξει η περίοδος του Ντέιτον και να ξεκινήσει για τη χώρα η ευρωπαϊκή της περίοδος. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Ε, μία πρόταση ψηφίσματο έχω λάβει για την όλη συζήτηση. Η συζήτηση λύγει τώρα και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Από τα μη γραμμένα μέλη υπάρχουν ε, ορισμοί σε επιτροπές ε, τροπών Περεκόβας, ε, Επιτροπή Ήτρε, που είναι μέρο των σχέσεων με την Αραβική Χερσόνησο. Αν δεν υπάρχουν σχόλια πάνω σε αυτό όταν εγκριθούν τα πρακτικά, αυτός ο ορισμός θα έχει θεωρηθεί εγκριθής. Ολοκληρώνεται εδώ αυτό το τμήμα της συνεδρίασης, η οποία διακόπτεται μέχρι τις 9 το βράδυ απόψε.